So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich begrüße... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά. Έχετε λάβει την σημερινή ημερήσια διάταξη. Υπάρχει καμιά επιθυμία για τροποποίηση, από ό,τι βλέπω όχι. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών. Γνωρίζετε πώς κάνουμε συνήθως, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Το ίδιο λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα. Φτάνουμε στο σημείο 3. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι ε, μεταδίδεται η σημερινή συνεδρίαση ζωντανά στο διαδίκτυο. Οι ακροατές ε, λοιπόν μπορούν να ακούσουν όλες σας τις παρεμβάσεις ε, και να δούνε και τη συμπεριφορά σας. Προσέξτε λοιπόν ε, και επίσης καλωσορίζω και τους ακροατές μας και προχωρώ στις ανακοινώσεις μου. Καταρχάς, Δεν έχουμε λάβει ακόμα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την διπλή χρήση προϊόντων. Αυτό με δυσαρεστεί, διότι το 2013 ήδη είχαμε συμφωνήσει οι τεχνολογίες ε, παρακολούθησης ε, να συμπεριληφθούν ε, στα προϊόντα διπλής χρήσης. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, προϊόντα που προορίζονται για βασανισμό ή για τα άλλα προϊόντα διπλής χρήσης να μην έχουμε εξυγχρονισμένη νομοθεσία. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω απέναντι στην Κομισιόν ότι τους παρακαλώ σύντομα να υποβάλουν σχετική πρόταση. Αυτό θα το πούμε γραπτός και στην Επίτροπο. Δεύτερη παρατήρηση που έχει να κάνει με τις προτάσεις νομοθεσίας της Κομισιόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι στις 10 Δεκεμβρίου Ε, εκπνέει το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ε, έχουμε συζητήσει πολύ καιρό ε, το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο και έχουμε υποβάλει και ψήφισμα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα νομοθετική πρόταση σχετικά με το πώς θα χειριστούμε χώρες ή περιφέρειες που ε, δεν χρησιμοποιούν τις ε, αρχές της ε, αγοράς στην τιμολόγησή τους. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλώ την Κομισιόν όσο γίνεται πιο σύντομα να υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση. Διότι εμείς ως Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε χρόνο για τις διαβουλεύσεις μας και για να ανταποκριθούμε στα δημοκρα... στις δημοκρατικές μας υποχρεώσεις. και θα θέλαμε να υιοθετήσουμε σχετική νομοθεσία πριν τις 11 Δεκεμβρίου. Και εδώ λοιπόν υποχρεούται η Κομισιόν να υποβάλει πρόταση. Και για αυτό το θέμα θα στείλω επιστολή στην Επίτροπο. Για να της εξηγήσω και την ανάγκη που υπάρχει για γρήγορη νομοθεσία στην περίπτωση αυτή. Θα ήθελα κατόπιν να σας θυμίσω ότι η Κένια την ημέρα μετά την επίσκεψη εδώ στην Επιτροπή μας υπέγραψε και στις 20 Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο της ε, Κένιας επικύρωσε την ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ε, με την Κένια μεταξύ Κένια και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι λοιπόν πληρεί η Κένια πια τι προϋποθέσεις. Γι' αυτό η έξι κατοξιδότηση πράξη που υπέβαλε η Κομισιόν είναι πλέον άνευ αντικειμένου. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν μπορεί να μου το επιβεβαιώσει αυτό. Αλλά υποθέτω πως ναι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την ε, απόσυρση αυτών των κατεξουσιοδότηση πράξεων, λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους. Παρακαλώ, ο Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, εξηγήσεις που μας δώσατε και όσον αφορά την Κίνα και όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξεις που αφαιρούν χώρες της Αφρικής. Διότι καταρχάς νομίζω ότι η προθεσμία 10 με 11 Δεκεμβρίου είναι αδύνατο να τηρηθεί διότι στην Μπρατισλάβα δεν ακολουθήθηκε η κατεύθυνση αυτή. Ακόμα λοιπόν και αν μέσα ή τέλη Οκτωβρίου λάβουμε σχετική πρόταση, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσουμε την προθεσμία. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε συζήτηση σχετικά με το πώς θα χειριστούμε το θέμα αυτό για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ε, δεύτερον, όσον αφορά τις κατεξουδότηση πράξης, ε, η Κομισιόν κατά την προηγούμενη ε, συνεδρίαση ανακοίνωσε την απόσυρση πέντε, νομοθετικών, πέντε πράξεων. Και συμφωνώ ε, με αυτά που είπατε. Στην Κένια είχαμε αφήσει ανοιχτό το θέμα αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε επιβεβαίωση από την Κομισιόν σχετικά με το αν έχουν αποσυρθεί οι προτάσεις αυτές, διότι είναι σημαντικό αυτό στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανατολικής Αφρικής. Sandra Galina kommt heute und ich werde sie dann Η Σάντρα Καλίνα θα έρθει εδώ σήμερα και θα τη ρωτήσω προσωπικά. Ο Χέλμουτ Σόλς αναφέρθηκε ήδη στο τελευταίο θέμα των ε, ανακοινώσεών μου, την ε, άτυπη συνάντηση στην Πρατισλάβα των Υπουργών Εμπορίου. Και Τρία θέματα συζητήσαμε εκεί μαζί τους. Και πράγματι, Χέλμουτ, το ένα θέμα ήταν τα εμπορικά εργαλεία σε σχέση με την Κίνα και την προσχώρησή της στον ΠΟΕ. Το, το Συμβούλιο συνεχίζει να έχει πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ανάγκη για μέτρα σε σχέση με την Κίνα. καθώς και όσον αφορά την τακτική διαδικασία, την, το πότε θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόταση. Το Κοινοβούλιο θα ήθελε σχετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν. και δεν επιτρέπεται συγκεκριμένες χώρες να εμποδίζουν τη διαδικασία αυτή. Και γι' αυτό, όπως σας είπα, θα ζητήσουμε από την Κομισιό να πάρει θέση στο θέμα αυτό. Δεύτερον, συζητήθηκε το θέμα των διαπραγματεύσεων TTIP. μεταξύ των κρατών μελών υπήρχαν πολύ διαφορετικές απόψεις. Ένα κράτο μέλο είπε ότι εφόσον δεν υπήρξε αποτέλεσμα υπό την κυβέρνηση Ομπάμα δεν θα είναι δυνατόν να συναυτεί η συμφωνία και γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις. Άλλοι είχαν ανάλογη θέση, αλλά είπαν ότι δεν θα πούμε να σταματήσουμε, αλλά θα σκεφτούμε μήπως κάνουμε νέα αρχή με νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως υπήρχε συνένεση ότι... Κανείς δεν θεωρεί πια ότι θα προλάβουμε με την κυβέρνηση Ομπάμα να διαμορφώσουμε παρκώς μια συμφωνία. Υποθέτω λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι τεχνικές συζητήσεις, όχι όμως πια με το στόχο να επιτευχθεί συμφωνία. Και τρίτον, είχαμε την συμφωνία ΣΥΤΑ. Μάλιστα, η Υπουργό Εμπορίου του Καναδά ήταν παρούσα και μας παρουσίασε τα συμφέροντα του Καναδά, που είναι από τους πιο στενούς εμπορικούς εταίρους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε από το 76 και μετά εμπορική συμφωνία η οποία ισχύει ακόμα. Έχουμε και 36 επιμέρους συμφωνίες καθώς και ε, κοινέ ε, πολιτικές δραστηριότητες. Η νέα καναδική κυβέρνηση λοιπόν επιθυμεί στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που εξέφρασε ο Υπουργός. είχα την αίσθηση ότι και 28 Υπουργοί Εμπορίου επιθυμούν στις 28 Οκτωβρίου να υπογραφεί η συμφωνία ώστε να, ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις. Υπάρχουν κάποιες μικρές επιφυλάξεις κάποιων κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη είπαν ότι θέλουν μια νομικά δεσμευτική δήλωση σχετικά με την ερμηνεία κάποιων σημείων της συμφωνίας. Καθώς και για τομείς που παραμένουν ανοιχτοί η Ρουμανία και η Βουλγαρία αναφέρθηκαν στην απελευθέρωση αποθεωρήσεις για τους πολίτες Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Έχω την εντύπωση όταν, ότι όταν δοθεί σαφές μήνυμα προς τους Καναδούς σχετικά με την υπογραφή, ε, οι Καναδοί θα αναλάβουν ε, βήματα σχετικά με την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις. Επίσης, συζητήθηκε το πεδίο εφαρμογής ε, της συμφωνίας. Είναι αδιαφεσβήτητο ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πει ναι, τότε ε, θα εφαρμοστεί προσωρινά μεγάλο μέρος της συμφωνίας. Φαίνεται να υπάρχει η κατανόηση ότι όσον αφορά το δικαστήριο επενδύσεων αυτό θα ε, ε, εξαιρεθεί καθώς ε, και μέρη του κεφαλαίου για τις υπηρεσίες, καθώς ε, και μέρη του κεφαλαίου για την πνευματική ιδιοκτησία όταν έχει ποινικέ συνέπειες, καθώς και κάποια ε, θέματα διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πει ναι, Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πει ναι, τότε ε, το 90% της συμφωνίας θα ισχύσει προσωρινά. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πολύ επικοδομητικό το άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, πιθανότατα θα υπάρξει στις 18 Οκτωβρίου δεύτερη άτυπη συνάντηση των Υπουργών, όπου θα ληφθεί επίσημα η απόφαση σχετικά με την υπογραφή για την ΣΥΤΑ. Και θα ξεκαθαριστεί το θέμα της απελευθέρωσης από θεωρήσεις, καθώς ε, και η επιπλέον κοινή δήλωση, καθώς ε, και η έκταση της προσωρινής εφαρμογής. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν επικοδομητική η συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου. Προσωπικά βρήκα και το κλίμα επικοδομητικό μετά από πολύ καιρό. Ε, διότι στα προηγούμενα συμβούλια δεν επικρατούσε τόσο ε, αρμονικό κλίμα. Ε, Χέλμουτ, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Μία ακόμα ερώτηση σχετικά με το TTIP. Είπατε ότι προφανώς θα, ε, θα ακολουθήσει την κατεύθυνση που είπατε, αλλά εγώ αναρωτιέμαι μήπως μια σαφής ε, εικόνα σχετικά με την εντολή που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχετικά με τις ε, δομές διαπραγμάτευσης. Θα ήταν σημαντικό και όσον αφορά την αντίδραση του κοινού. Εάν το Κοινοβούλιο να το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί αυτήν την, ε, ε, το διάστημα παγώματος, πώς θα το χειριστούμε. Πρόεδρος. Από άποψη ε, δεν είναι πολύ απλό το θέμα, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε. Σάντρα. Καλώς ήρθατε. Πριν λίγα λεπτά συζητούσαμε το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων για την Κένια. Στις 20 Σεπτεμβρίου η Κένια επικύρωσε την ε, Συμφωνία Εμπορικής Εταιρικής Σχέση και ήθελα να ρωτήσω αν έχουν αποσυρθεί οι προτάσεις. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Η Κομισιόν, λοιπόν, αποσύρει τις εξουσιοδότηση πράξη. Ε, σημείο 4. Πρωτού προχωρήσω στο σημείο 4, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα από την Γερμανία ε, της εταιρεία για τη διεθνή συνεργασία που ασχολείται με την παρακολούθηση των εμπορικών ε, εταιρικών σχέσεων. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά. Ακόμα και η Κομισιόν χαίρεται. Ωραία. Προχωράμε στο σημείο 4. Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το έτος 2007 οι συντονιστές το ενέκριναν. Ενημερωτικά λοιπόν. Σημείο 5. Κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Έναν τριμερή διάλογο έχουμε που συνεχίζεται και μάλιστα βρίσκεται στην ε, τελική του φάση. Ε, πρόκειται για τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Μιλάμε δηλαδή για την εφαρμογή αυτών που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό, τέσσερα συγκεκριμένα μέταλλα να φτάνουν από τα ορυχεία ε, στην κατανάλωση με τρόπο σωστό και λογικό στις 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε τεχνική συνάντηση και αν όλα πάνε καλά τότε στις 19 ε, Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί το θέμα ε, με τη βοήθεια του κυρίου Βίνκλερ που είναι ο εισηγητής μας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολύ σύντομα και θα σας ε, τονίσω το εξής. Τι έχω αξιολογήσει για την κατάσταση και επίσης θα σας πω και ένα αίτημά μου για τους σκιώδεις συζητητές συναδέλφους αλλά και για δύο από τους συντονιστές η εκτίμηση που έχω κάνει αφορά το ότι η γραμματεία μα έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για το θέμα και την ευχαριστούμε και θα συνεχίσει αυτή τη σκληρή δουλειά γιατί ακόμα δεν ολοκληρώθηκε το έργο τη γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σα ευχαριστούμε για όσα κάνατε και επίση. Το αίτημά μου προς συντονιστές και σκιώδες είναι, φυσικά αφού τους ευχαριστήσω για τα όσα έκανα και εκείνη, ότι θεωρώ πως θα δώσουν εντολές στους συνεργάτες μας, στους εμπειρογνώμονες, σε όλους όσοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις τεχνικές συναντήσεις που εξήγησε Πρόεδρε και επομένως οι συνεργάτες, προσωπικό και εκείνοι επομένως ε, να μπορέσουν να μετάξουν στις συναντήσεις σε αυτό το πνεύμα της πολιτικής συμφωνίας και επίσης όλοι να ξέρουν ότι κινούμαστε στο μήκο κύματο του συμβασμού όλοι, όλοι αυτό θέλουμε στο κοινοβούλιο ήρθε τώρα η ώρα να κλείσουμε το θέμα και να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό νομοθέτημα ο πρόεδρος Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ Σας ευχαριστώ για τον ενεργό ρόλο που έχετε παίξει σε όλη αυτή τη διαδικασία και πράγματι, όπως είπατε, θα έχουμε ένα σημαντικό πακέτο νομοθεσίας ε, και ένα ορόσημο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έχει πετύχει δεσμευτική νομοθεσία σχετικά με την χρήση ε, ορυκτών. Θα είναι ένα πρώτο βήμα όσον αφορά τις εμπορικές αλυσίδες σε όλο τον κόσμο, είτε μιλάμε για ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, είτε μιλάμε για υφάσματα και ε, είδη ένδυσης. Ευχαριστώ πολύ και έτσι φτάνουμε στο σημείο 6 της ημερησίας διάταξης που συνδέεται κάπως με το θέμα αυτό. Δηλαδή, τι ισχύει όσον αφορά την εφαρμογή των εργασιακών προτύπων ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Όσον αφορά την βιωσιμότητα, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των εργασιακών προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Και αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει και με την συμφωνία με τον Καναδά, αλλά συνδέεται και με πολλά άλλα θέματα την Κολομβία, το Περού, το Μπαγκλατές, ε, τις ε, Φιλιππίνες, ε, που νομίζω είναι επίσης πολύ επίκαιρο θέμα. διότι προβλέπεται να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις για, εμπορικές, για εμπορική συμφωνία, αλλά οι, οι εξελίξεις στις Φιλιππίνες δεν υπόσχονται πολλά καλά. αλλά και με το Βιετνάμ έχουμε συνάψει συμφωνία εμπορική, αλλά το θέμα των συνδικαλιστικών ε, δικαιωμάτων ε, βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και με την Νότια Κορέα έχουμε το και πέντε χρόνια σχετική συμφωνία. αλλά η παράγραφος ε, κατά των απεργιών δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να ακούσουμε τη θέση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το θέμα αυτό. Επίσης, τίθεται το θέμα της ε, αξιοπρεπούς εργασίας ε, στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Είναι λοιπόν θέματα αυτά που συζητάμε εδώ στην Επιτροπή μας. Η κυρία Κορίν Βάγκα, Διευθύντρια του Τμήματος για τα Διεθνή Πρότυπα στη, στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, βρίσκεται μαζί μας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής που καλέσετε τον ILO για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εμείς εκτιμούμε την ευκαιρία αυτή. Ώστε να συζητήσουμε τα πρότυπα αυτά σε έναν αριθμό από χώρες. Ε, να ρωτήσω, Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω για την παρέμβασή μου. Ίσως 10 με 15 λεπτά, λέει ο Πρόεδρος. Το επόμενο σημείο είναι για τις 4. Μάλιστα. Καλό που ρώτησα, λοιπόν. Άρα δεν θα μπορέσω να καλύψω όλες τις χώρες για τις οποίες ενδιαφέρεστε, αλλά μόνο κάποιες επιλεγμένες υπό το φως της πρόσφατης ε, συζήτησης τον Ιούνιο στη Γενέβη. Η επιλογή αυτή έγινε ε, επί τη βάση του ενδιαφέροντός σας και θα τις διατρέξω αλφαβητικά. Παρακαλώ μην διαβάσετε καμία άλλη σημασία σε αυτή τη σειρά. Και ξεκινάω από τον Μπαγκλαντές λοιπόν. Και πάλι εφέτος προσεκλήθη για την Επιτροπή της ε, Επιβολής των Προτύπων για τη Σύμβαση 87 για την ελεύθερη εγκατάσταση, μάλλον για την, ε, τον ελεύθερο συνεταιρισμό. Τα συζητήματα που συζητήθηκαν ήταν παραβίαση των ε, αστικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών ενώσεων, νομικών εμποδίων για την καταχώρηση των εταιριών, απουσία μηχανισμού καταπολέμησης ε, πρακτικών κατά του ελεύθερου εμπορίου, όπως και διαδικασίες σχετικά με τις εξαγωγές, τις ζώνες εξαγωγής μάλλον. Η Επιτροπή του Συνεδρίου σημείωσε με ικανοποίηση ότι σε σχέση με την ελευθερία του συνεταιρίζεστε πρότεινε στην κυβέρνηση την ανάλυση διαφόρων μέτρων συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του τελευταίου νομοθετήματος που είχε υποβληθεί σχετικά με αυτό να ερευνήσει όλες τις διακρίσεις κατά των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιταχυνθούν διαδικασίες καταχώρησης των ευρωπαϊκών εταιριών όπως και να υλοποιηθούν οι συστάσεις της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου που επισκέφθηκε τον Απρίλιο φέτος από τους δύο αντιπροέδρους της Επιτροπής της Επιβολής των Προτύπων. Ίσως να σας να ξέρετε ότι ο ΑΕΛΟ προσεκλήθη μόλις σε μια ακρόαση του Κοινοβουλίου Τετάρτη και Πέμπτη και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί νέα νομοθέτηση νέα νομοθετική πρόταση για τις εξαγωγικές ζώνες ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα συνδεδεμένα κεφάλαια και τις ε, σχετικές επιθεωρήσεις εργασίας. Να σας δώσω τώρα μια επικαιροποίηση για το που βρισκόμαστε σχετικά με τη συμμόρφωση για τη σύμβαση των επιθεωρήσεων εργασίας που θα θυμάστε ότι είχε συζητηθεί στην ε, Επιτροπή Συνεδρίου μετά το επεισόδιο της ε, Πλάζα σχετικά με ε, κάποια προβλήματα που είχε σημειώσει η, ομάδα επιθεώρησης εργασίας και κενά στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά και με την επιβολή και τον έλεγχο, ε, σημειώθηκε κάποια πρόοδος γιατί όπως θα γνωρίζετε έχουμε ένα πολύ μεγάλη κλίμακα σε ε, πρόγραμμα ενίσχυσης, σε συνεργασία, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι. Ε, το Σεπτέμβριο πέρυσι υιοθετήθηκε το νομοθέτημα σχετικά με την ε, ελεύθερη αγορά όπως και με τις επιθεωρήσεις ασφάλειας κατά της πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων στα κτίρια. Σε σχέση λοιπόν με κάποια από αυτά τα θέματα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο παρότι όπως γνωρίζετε είμαι βέβαιη ε, παραμένουν διάφορα προβλήματα και προκλήσεις. Αλλά έχουμε κινήσει ξεκάθαρα τη διαδικασία και αυτή προχωρεί. Να περάσω στο Εκουαδόρ Το Εκουαδόρ προσεκλήθη για μη συμμόρφωση της ε, σύμβασης για τις συλλογικέ συμβάσεις εργασία. Το πρωταρχικό θέμα ήταν η άρνηση δικαιωμάτων συλλογικών συμβάσεων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και ο αποκλεισμό του δημόσιου τομέα προεκτάθη το Δεκέμβριο πέρυσι με συνταγματική τροποποίηση στη χώρα αυτή είναι σημαντικό να γνωρίζετε ε, ότι φέτος το Σεπτέμβριο προτάθηκε από την Συνομοσπονδία των ε, Συνδικαλιστικών Ενώσεων των χωρών της Αμερικής και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας μετά τις εξελίξεις του Αυγούστου από τις ενώσεις των διδασκόντων, των διδασκάλων ελάβαμε από τον τύπο την απάντηση του Υπουργού του Αρμόδιου, ο οποίος υποστηρίζεται ότι η σχετική καταγγελία προέρχεται από, όχι από συνεργαστική ένωση, αλλά από άλλο φορέα της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό το παρακολουθούμε στενά. Επίσης, η αντιπροσωπεία που προσήλθε δεν ήταν τριμερής, δυστυχώς. Ε, σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα ζητήσαμε εξηγήσει από την κυβέρνηση και θα το συζητήσουν οι εμπειρογνώμονες ε, Νοέμβριο και Δεκέμβριο φέτος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση στο Εκουαδόρ. Για την Κορέα, πρόεδρε, ίσως να σας ενδιαφέρει να ξέρετε τι συνέβη. Εντεφέτος δεν συζητήσαμε την Κορέα, την συζητήσαμε πέρυσι αυτό που υπόθηκε σε σχέση με την σύμβαση ε, κατά των διακρίσεων, διακρίσεων που προκύπτουν κυρίως από ανισότητες ε, στην ε, αγορά εργασίας και στην ελεύθερη πολιτική έκφραση άποψη των διδασκάλων. Η κυβέρνηση είχε αναλάβει διάφορα νομοθετικά μέτρα μετά τη συζήτηση που είχε γίνει τότε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων επανεξέτασε το υλικό που υπέβαλε η κυβέρνηση της Κορέας σχετικά με τα νομοθετικά αυτά μέτρα από τη συζήτηση του Ιουνίου του 2015 δηλαδή και μετά αυτό που σημείωσαν οι εμπειρογνώμονες ήταν το γεγονός ότι οπωσδήποτε οι διδάσκαλοι ε, υποβάλλονται σε διοικητικά, διοικητικές κυρώσεις λόγω της συμμετοχής τους σε πολιτικές ε, δραστηριότητες. Ίσως επίσης να σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι ότι follow-up της συζήτησης και της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων, ο ILO υποστηρίζει την κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξετάσουμε ποια είναι τα υπόλοιπα νομοθετικά κενά για την Σύμβαση 111. Αυτή που σας έλεγα πριν. Μιλώντας για την Κορέα επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΟ εξέφρασε νέες ανησυχίες σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι και ο πρόεδρος της ε, Ομοσπονδίας Συνδικάτων της Κορέας ε, καταδικάστηκε σε πέντε έτη σχετικά με παράνομες δραστηριότητες μαζί με 19 εκπροσώπους τον Νοέμβριο πέρσι. Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν του ΑΕΛΟ αναφέρθηκε στην παρέμβασή του γιατί πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα ότι προβλήματα που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν επανέρχονται στο προσκήνιο. Υπάρχει και μια πρόθεση απεργίας αυτή την εβδομάδα και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην Κορέα σχετικά με αυτό. Τώρα, για την Μιανμάρ, η οποία δεν συζητήθηκε όπως ίσως να ξέρετε στο συνεδρίο, αλλά μου είπαν ότι σας ενδιαφέρει να παρακολουθείτε το θέμα αυτό. Τρεις βασικές περιοχές παρεμβάσεως χρειάζονται ώστε η Μιανμάρ να προχωρήσει στο επίπεδο συμμόρφωσης ε, για το κράτος δικαίου και τα πρότυπα εργασίας. Υπάρχει βασική αναθεώρηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άμεση ανάγκη υποστήριξη των θεσμών που είναι υπεύθυνοι για την επιβολή και η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των φορέων της αγοράς εργασίας στη χώρα αυτή. Έχουμε κινήσει ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση της Μιανμάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τον ΑΕΛΟ τον Νοέμβριο 14 και από το Μάρτιο του 2015 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υποστηριχθεί η Μιανμάρ σε αυτές τις τρεις περιοχές. Με λοιπόν την ενίσχυση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αυτήν την εβδομάδα το δεύτερο φόρουμ των ενδιαφερομένων φορέων διοργανώνεται προκειμένου να συζητηθεί η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και η ε, θεσμική ικανότητα που χρειάζεται για να ε, εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Όλα αυτά τρέχουν και χάρη στην ε, υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Έχουμε δει κάποιες πρόοδους, αλλά βεβαίως πολλά μένει να γίνουν έχει γίνει κάποια πρόοδος σχετικά με την επικαιροποίηση κάποιων σημαντικών τμήματων της νομοθεσίας. Κοιτάω και το ρολόι μου, λέει η ομιλητρία. Και φαντάζομαι ότι μπορώ ακόμα να πω δύο λόγια και για τις ε, Φιλιππίνες και για την αλυσίδα προμήθειας εκεί. Για τις Φιλιππίνες λοιπόν. Ήταν μία από τις χώρες που συζητήθηκαν στην Επιτροπή ε, ε, συνεδρίου για την Σύμβαση 87 είχαμε κάποιες πρόοδους σχετικά με τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού για τις παραβιάσεις μεταξύ άλλων και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει πρόοδος, και αυτό σημειώνεται, στην, έρευνα διαφόρων κρουσμάτων ε, βίας κατά της Ένωσης Έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα από τις επαρκείς έρευνες σχετικά με εγκληματικές ε, πράξεις όπως δολοφονίες ε, κατά μελών συνδικαλιστικών ενώσεων και την υποδοχή μιας ε, αποστολής ακριβώς με το θέμα αυτό έκτοτε ήμασταν σε θέση να προχωρήσουμε μια συζήτηση με την κυβέρνηση για να έχουμε μια αποστολή άμεση επαφής ε, ε, του χρόνου για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά τα θέματα. Έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις, η δέσμευση όμως της κυβέρνησης ε, εξακολουθεί να υφίσταται με τον ΑΕΛΟ για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα θέματα που σημείωσε η Επιτροπή Συνεδρίου. Τέλος, για την ε, παγκόσμια λυσίδα προμήθειας. Υπήρξε μια περίπλοκη και μακροσκελή συζήτηση για το σημαντικό θέμα αυτό φέτος τον Ιούνιο. Ε, το Παγκόσμιο Συνέδριο Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία της ε, προμήθειας. Περίπλοκες, όπως έλεγα, και μακροσκελή συζητήσει. δύσκολα, δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα. Εξήχθησαν κάποια, και η συζήτηση και τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την πολυεπίπεδη φύση των αλυσίδων προμήθειας, την συνεισφορά τους ε, στην παγκόσμια ανάπτυξη της οικονομίας και τις ε, σχετιζόμενες ε, ελλείψεις που έχουμε στις συνθήκες εργασίας έχουμε μια σειρά από συμπεράσματα για δράση πρέπει να αναλυθεί από κυβερνητικού φορείς, από τις εταιρείε και από τους κοινωνικούς εταίρους. Στις 22, 23 και 25 παραγράφου των συμπερασμάτων ιδιαίτερα παρέχονται σαφεί οδηγίες στον ΆΕΛΟ για περαιτέρω δράσεις και αν ε, διαβάσετε την παράγραφο 23 που εγώ δεν το κάνω εδώ λέει ομιλήτρια Εδώ έχουμε μια σαφής περιγραφή των όσων καλεί το Α.Ε.Λ.Ο να παρακολουθήσει, ένα πρόγραμμα δράσης δηλαδή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο ILO χρησιμοποιεί το σύνολο της εμπειρογνωμοσύνης του, της εμπειρίας του, της δυνατότητάς του να διοργανώνει ε, συναντήσεις και να διαφωνούν το διάλογο Και έχουμε πέντε άξονες για την ανάπτυξη του σχετικού αυτού προγράμματος, ε, γνώση και διάχυση, ανάπτυξη δυναμικού για όλους τους φορείς που σχετίζονται με την ε, αλυσίδα προμήθειας. Επίσης, όπως αναφέρετε και εσείς νωρίτερα, Πρόεδρε, ε, φορείς υποστήριξης και προώθησης της αξιοπρεπούς εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις και για άλλες βασικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, ε, συμβουλές και υποστήριξη στον ILO και εταιρικέ σχέσεις, τέλος. Γιατί κανείς δεν μπορεί να επιτύχει βιώσιμες ε, μεταρρυθμίσεις ε, χωρίς πολυμερή στήριξη. Ένα πρόγραμμα δράσης θα υποβληθεί λοιπόν ή στο Διοικητικό Σώμα του ΑΕΛΟ τον Νοέμβριο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσει θα εξαχθούν στο σώμα αυτό και τι οδηγίε θα δώσει το σώμα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματο δράση. Οπωσδήποτε όμω, έχουμε ήδη την οδηγία να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην παρέμβασή μα. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό ήταν μια σύντομη ενημέρωση. Update. Σας ευχαριστώ για την σύντομη αυτή ε, ε, ενημέρωση. Θα δώσω το λόγο τώρα ε, στους ευρωβουλευτές ε, για δύο λεπτά το πολύ ο καθένας. Κυρία Μινές, παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Βάργα. Και επίσης πρέπει να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενημέρωση που αφορούσε τόσες χώρες, αλλά έχουμε και άλλες χώρες οι οποίες ακόμα προσκρίνουν σε κάθε δυσκολίες σε σχέση με αυτές τις βασικές ελευθερίες που προβλέπει ο ΆΕΛΟ πιστεύω ότι το κείμενο της συνθήκης ενθαρρύνει στο να προσυπογραφούν και άλλες ε, θεμελιώδεις συνθήκες αλλά δεν προβλέπεται καμία κύρωση για τις χώρες που ακόμη δεν τις έχουν προσυπογράψει. Οπότε για πέστε μας τι γίνεται, τι εξελίξεις έχουμε τώρα όσον αυτό το πρόγραμμα εργασίας για την ΣΕΤΑ. Επίσης για πέστε μας τη γνώμη σας όσον αφορά το συμπληρωματικό πρωτόκολλο και ιδίω πέραστε μα, η γίνεται όσον αφορά τι συνθήκες εργασίας. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Τι πρεσβεύει από αυτού ο Άγγελο, ο επόμενος. Ο κύριος Σόλτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βάγκα για την ε, σύντομη αλλά πολύ σαφή παρουσίασή της. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή στην Γενέβη για δεσμευτική συμφωνία του ΟΗΕ σχετικά με την ευθύνη των ε, επιχειρήσεων. Σε τι βαθμό συμμετέχει εδώ η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και σε τι βαθμό ενδιαφέρεται για την εφαρμογή της, διότι νομίζω ότι το θέμα των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα που θα πρέπει να διασφαλίσουμε οριζοντίως σε σε όλες ε, τις ε, συμφωνίες κλπ. Αλλά η ερώτησή μου είναι σε τι βαθμό πράγματι συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες. Και μία δεύτερη ερώτηση. Ε, πώς πραγματοποιείται η επιλογή των ανθρώπων που κάνουν την παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και την ομιλήτρια. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την πολιτική για το TRIPS, όπως ξέρετε, έχουμε το, το κεφάλαιο για την βιωσιμότητα και πάντοτε οι σοσιαλδημοκράτες θέλουν να προχωρήσουν προς τα εκεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όσον αφορά τα πρότυπα εργασία για αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε τις σχετικές ε, συμφωνίες τελευταία, δηλαδή πανεπιστημιακή, ε, έχουν αξιολογήσει το ότι δεν υπάρχει πρόοδο σε αυτό το μέτωπο. Για πετε μου τις σκέψεις. Επίσης, για άλλες δύο χώρες θέλω να ρωτήσω για την Κορέα συμφωνώ με όσα είπατε και ανησυχούμε ότι έχουν πάρει την κάτι τα, τα εργασιακά δικαιώματα δεν έχει κυρώσει την ε, Σύμβαση 98 τι λέτε, τι μπορεί να κάνει για να βελτιωθούν τα πράγματα τέλος κάτι άλλο που δεν προφτάσετε να μας πείτε για την Τουρκία λένε από το 90 ότι κάπως τα πράγματα βελτιώνονται όσο πρέπει την εργασία των ανηλίκων, αλλά από τότε που φούντωσε το προσφυγικό, τα πρά... η τάση είχε αντιστραφεί. Έχετε, διατηρείτε επαφές τέλο πάντων, συγχύσετε επαφές με την Τουρκία πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ. Σάντσες. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ θέλω να ρωτήσω για την εμπορική πολιτική της Ένωσης και συγκεκριμένα όσον αφορά την ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Για να μας πει ΑΕΛΟ η κοινωνική ρήτρα ε, έχει αρκετή δεσμευτικότητα. Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για κυρώσεις. Αν χρειαστεί. Δεύτερη ερώτηση. Θεωρείται ότι επαρκεί μια τέτοια εμπορική συνθήκη για να έχουμε τέτοιες ρήτρες, γιατί υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της ερμηνείας του ΑΕΛΟ και των οργάνων που προβλέπονται για την εφαρμογή του ΣΕΤΑ. Ο επόμενος. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε πολύ ε, χρόνος, ε, αλλά είπατε για την ε, Κορέα ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Εδώ και πέντε χρόνια όμως έχουμε και συμφωνία εμπορική με την Κορέα, στην οποία η Κορέα δεσμεύεται να εφαρμόσει και να επικυρώσει τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Βρίσκεται ότι ε, υπάρχει ε, επαρκής πίεση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αλλιώς τι να τις κάνουμε τις εμπορικές συμφωνίες εάν δεν ασχολείται κανείς μετά. Ερωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει στηρίξει επαρκώς για να ασκηθεί πίεση στην ε, κυβέρνηση της Κορέας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εκπρόσωπο του ΑΕΛΟ για ε, την ε, σημαντική της εισήγηση πριν υποβάλουν ερώτηση μου να τονίσω ότι στις 5 Ιουλίου το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα. Ε, ε, η συγκήτρια από ότι ακριβώς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είναι τα κεφάλαια για την βιώσιμη ανάπτυξη ε, πιο ουσιαστικά, πιο συνεπή. Ε, λογικά σε σχέση με τα δικαιώματα και τα πρώτη εργασία θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να γίνει σχετική κύρωση όσον αφορά τις 8 επιμέρους ε, συμφωνίες. Ε, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και επίσης εσείς έχετε την παγκόσμια διαχείριση των Global Supply Chains και επίσης θα πρέπει η προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων είναι ένα βασικό θέμα για το Κοινοβούλιο όσον αφορά την συνεργασία μας με τον ΑΕΛΟ. Επίσης συμφωνώ με αυτά τα οποία ρώτησαν οι συνάδελφοι όσον αφορά την ε, ΣΕΤΑ αλλά και τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη διότι το ότι συνεχίζουμε να έχουμε απλώς σε επίπεδο ενδείξεων ε, τις συνθήκες εργασίας χωρίς να υπάρχει κάποιο δεσμευτική ρύθμιση και επομένω είναι θέμα κύρωση των ε, συνθηκών με τον ILO. Οπότε θα πρέπει να εξετάσει την ΣΕΤΑ ο ILO αλλά και την συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Επίσης θα ήθελα να ακούσω από εσά τι ισχύει για την Τουρκία γιατί ακριβώς έχουμε εκεί το ζήτημα της εργασίας των ανηλίκων. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αγνοήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ενέργειες μπορείτε να αναλάβετε επίσης, τι γίνεται και με τον Μπαγκλαντές όσον αφορά την τήρηση της σχετικής συμφωνίας με την χώρα εκείνη. Τελευταία αλλά σημαντική εσείς, συνάδελφοι, και εγώ να ευχαριστήσω την ε, ε, ε του ΑΕΛΟ για το έργο που επιτελεί. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι το ότι εμείς αποδίδουμε την έμφαση στις εμπορικές συμφωνίες που εκάστοτε όλο ένα και με περισσότερες λεπτομέρειες υπογράφουμε ε, για τα εργασιακά δικαιώματα και λοιπά και για την αηφορία υπό την ηγίδα του ΑΕΛΟ. Όμως για πέστε μου, τι γίνεται άμα έχει υπογράψει μια χώρα, μια σύμβαση, μια συνθήκη και κατόπιν ε, κάνει κάποιες... Ε, τέλο πάντων κάποιο δίκαιο, κάποια νομοθετήματα που δεν συνάδουν προς την συνθήκη που έχει υπογραφεί. Τι προβλέπετε επίσης, θα ήθελα να μας ενημερώσετε κάπως περισσότερο να γίνεται όσον αφορά τις Φιλιππίνες, διότι πρόκειται να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό στο Κοινοβούλιο να είμαστε ενδελεχώς ενημερωμένοι για την πραγματική κατάσταση. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα για να δούμε πώς θα βαδίσουμε προς την σύνοψη αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σάντρα, έχεις τρία λεπτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των προτύπων του ΆΕΛΟ, ιδίω για την Νότια Κορέα. Um, Ευχαριστούμε που μας καλέσατε και εμείς ε, έχουμε τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση που συνεργάζεται με τον ΑΕΛΟ αλλά και την Γενική Διεύθυνση για την Εμπορική Πολιτική που ασχολείται με τις ε, συμφωνίες ε, που έχουν συναυθεί, θα συναυτούν με τις εν λόγω χώρες, οπότε είναι συνεχή συνεργασία μας με τον ΑΕΛΟ και με την ευκαιρία αυτή δημοσία να ευχαριστήσω για τα όσα επιτελούν. Βεβαίω και δημιουργούν ανησυχία ε, κάποια αυτά που ακούσαμε ε, τι να σας πω, να, να, να σας απαντήσω τηλεγραφικά και μετά να τα συζητήσουμε για τον Μπαγκλαντές. Όχι, δεν έχουμε ε, αφετηρία τη συμφωνία με τη χώρα, αλλά έχουμε ως αφετηρία επαφών μας με το σύστημα γεμμένων προτιμήσεων και όσον αφορά την Κορέα. Είπαμε ότι υπ' αυτής της βάσεως θέλει να κάτσει στο τραπέζι ο ΑΕΛΟ. Αλλιώς ο ΑΕΛΟ θα βγει έξω από το παιχνίδι. Επίσης έχουμε και κάποιες άλλες χώρες που αναφέρθηκαν ας πούμε για την Μιανμάρ και είπα αυτής της περιπτώσεως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την άμεση συμμετοχή σε κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πολύ βασικά όλα αυτά για μας, οπότε έχουμε επίσης και την Συμφωνία 111 για την ε, Κορέα. Άρα βρίσκεται εν εξελίξη η επεξεργασία αυτών των θεμάτων. Δεν συνεργαζόμαστε με όλα, με όλο το θεματολόγιο, αλλά τέλος πάντων εμείς τι έχουμε επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπαμε ότι θέλουμε κάποια πρότυπα τα οποία στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε για την εμπορική μας πολιτική να στηρίξουμε τον ΑΕΛΟ, τη βασική συνθήκη, τη βασική συμφωνία και για τα πρότυπα. Ε, ας ε, λάβουμε υπόψη και καμιά φορά τι ισχύει στην Ευρώπη. Αυτό λέω εγώ στους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Επίσης ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που δώσατε στον ΑΕΛΟ να έρθει εδώ και να τοποθετηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν εδώ οι εταίροι μας να μας πούν τι γίνεται για τις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου κλπ. Και επίσης βεβαίως και είναι πολύτιμο το ψήφισμα της βουλευτού κυρίας ε, Φορέντζα και έτσι δείχνουμε στους εταίρους μας ότι προσέχουμε τα εργασιακά δικαιώματα επίσης. Ένα άλλο στοιχείο ενθουσιασμού είναι τις στρατηγικές εμπορικές πολιτικές. Πολύ σημαντικό αυτό γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την υλοποίηση των όσων προβλέπονται για τα εργασιακά δικαιώματα ή στις χώρες εκείνες για τις οποίες έχουμε συμφωνίες. Αλλά προσοχή, δεν θεωρούμε ότι το εμπόριο είναι η μόνη πολιτική, το μόνο εργαλείο. Γι' αυτό και έχουμε την υπηρεσία εξωτερική δράση. Έχουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μόνο τα εργασιακά πρότυπα. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλές οι ερωτήσεις που ακούσαμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ. Κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν σχετικές μεταξύ τους όσον αφορά τα πρότυπα ε, και τι ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Νομίζω ότι από πλευρά της Διεθνού υπάρχουν εδώ τρία σημαντικά θέματα. η σχέση των ε, ρητρών εργασίας, η συνάφειά τους ε, και η σωστή ε, χρήση τους και τα διεθνή πρότυπα εργασίας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Ανησυχεί όσον αφορά τις συμφωνίες που επιλέγουν τις πιο ευνοϊκές ρήτρε και δεν χρησιμοποιούν τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ως σημείο αναφοράς και ως ε, κύριο μέσο για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Για μας λοιπόν σημαντικό είναι αυτές οι εμπορικές συμφωνίες να παραπέμπουν στα κατάλληλα εργαλεία και να χρησιμοποιούν το σύστημα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ως ε, σύστημα για την ε, παρακολούθηση της συμμόρφωσης όσον αφορά το θέμα του κατά πόσο είναι αποτελεσματικές, αν είναι επαρκώς δεσμευτικές, ε, τι γίνεται με τις κυρώσεις. Εδώ δεν έχει πολλά να πει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Αυτό που βλέπουμε είναι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που να αποτελούν ε, μοχλό για την χρήση των ε, διεθνών προτύπων εργασίας. Η πείρα μας έχει δείξει ότι οι συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου αποτελούν ένα κίνητρο αλλά δεν αρκούν. Χρειάζεται ε, στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και έχουν την πολιτική βούληση να βελτιώσουν τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα εργασίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα το Βιετνάμ. Στο Βιετνάμ συμμετέχουμε εδώ και πάνω από μια δεκαετία για να τους βοηθήσουμε να συμμορφώνονται με τα εργασιακά πρότυπα και να τους βοηθήσουμε στη μετάβαση προς πιο προηγμένες ε, βιομηχανικές σχέσεις και εργασιακές σχέσεις. Όλα αυτά αποτελούν πολύ χρόνο. Θέλουμε λοιπόν επικοδομητική συνεργασία και δεν θέλω να μπω τώρα στο παιχνίδι να ευχαριστούμε ένα τον άλλον, αλλά η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί πολύ σημαντική υποστήριξη. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να συμμετέχουμε πολύ πιο ουσιαστικά. Όσον αφορά τον αντίκτυπο όλων αυτών, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ερωτήσεις, διότι είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει κανείς ε, στοιχεία. Προσπαθούμε να έχουμε επιστημονική ε, προσέγγιση στη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Τον ε, Νοέμβριο θα εκδοθεί έγγραφο σχετικά ακριβώς με αυτό το θέμα, με τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τα εργασιακά πρότυπα και τους διάφορους μηχανισμούς για την εφαρμογή των προτύπων αλλά βέβαια απομένει πολλή δουλειά να γίνει για να έχουμε ε, μια σωστή αξιολόγηση αντικτύπου. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι αυτό που εκτιμούμε περισσότερο είναι το να έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν χώρο για την προώθηση των εργασιακών προτύπων σε μια χώρα. Και βέβαια ακόμα και η αρχή πρόοδος είναι καλύτερη από ε, την έλλειψη πρόοδου. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιχειρήσεις, βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους συναδέλφους μας πάνω στο θέμα αυτό. Πρόκειται για μη δεσμευτικά μέσα που προσφέρουν όμως ένα δημιουργικό χώρο στον οποίο ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για να προωθήσει τα εργασιακά πρότυπα. Έχουμε λοιπόν συνεργασία πάνω στο θέμα αυτό και πώς επιλέγουμε τις χώρες. Υπάρχει μια σειρά κριτηρίων που ε, ε, χρησιμοποιούν οι δύο αντιπρόεδροι για την επιλογή των 24 χωρών κάθε χρόνο. Εξετάζουμε την μακροχρόνια μη συμμόρφωση, την σοβαρότητα των ε, παραβάσεων και την θέση της κυβέρνησης. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εργοδοτών και Εργαζομένων. Όσον αφορά το αν έχουμε διάλογο με την Κορέα υπό το φως της νέας επικύρωσης, ναι, έχουμε συνεχιζόμενο διάλογο, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για εξέταση της δυνατότητας να επικυρωθούν νέα μέσα. Και δεν έχουμε συνομιλίες όσον αφορά την Σύμβαση 98. Για την Τουρκία και την εργασία ανηλίκων ε, έχετε δίκιο, ε, σημειώνουμε βελτίωση και μέσω της τεχνικής βοήθειας Ε, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη όσον αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι η προσφυγική κρίση σημαίνει ότι έχουν ε, προσέλθει στην ε, Τουρκία πάρα πολλοί ανήλικοι που χρησιμοποιούνται μετά στην εργασία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη, τεχνική βοήθεια για να μην χάσουμε ε, τα όσα έχουμε κερδίσει στην Τουρκία όσον αφορά την ε, εργασία ανηλίκων. Όσον αφορά τις Φιλιππίνες, πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν ως εξής. Ε, κάποια νομοσχέδια δεν πέρασαν από το Κοινοβούλιο, αλλά η υιοθέτηση της νομοθεσίας αυτής ε, αποτελεί προτεραιότητα για την ε, επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Επίσης ε, προβλέπεται αποστολή αρχές του επόμενου έτους όπου θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση όσον αφορά τα θέματα αυτά και επίσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για το Εμπόριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορέσουμε να παράσχουμε βοήθεια σε θεσμούς που προωθούν ε, τον κοινωνικό διάλογο. Ελπίζω λοιπόν ε, κύριε Πρόεδρε να μπόρεσα να απαντήσω στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βάρκα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω θα είμαστε σε επαφή για να βελτιώσουμε τα εργασιακά πρότυπα για ε, τους ανθρώπους ε, σε όλο τον κόσμο. Προχωράμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7. Πρόκειται για την πρώτη ψηφοφορία της έκθεσης ε, για την ρήτρα διασφάλισης της Συμφωνίας Κολομβίας και Περού. Η συγκίτρια είναι η κυρία Desarnes. Και χρειαζόμαστε τις κάρτες σας για την τελική ψηφοφορία. Γι' αυτό ο συνήθως ε, θα κάνουμε και μία δοκιμή πρώτα. Αρχή λοιπόν της ε, δοκιμαστικής ψηφοφορίας. Ωραία, ολοκληρώθηκε. Όλα λειτουργούν έξοχα και εκπροσωπούνται σωστά οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Προχάμε λοιπόν στο σημείο 7. Ρήτρα διασφάλισης ε, για τις μπανάνες. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 20, δεύτερο τμήμα, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Compromise 4. 4. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 δεύτερο τμήμα. 35 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις, ε, τροπολογία 14, υπέρ, κατά, Άποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση της 16, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τροπολογία 15. Ηλεκτρονική επαλήθευση αρχής ψηφοφορίας. Äh, Abstimmung geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το νομοθετικό ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θα ήθελε η συγγήτρια να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ε, προτείνω, μια και έχουμε πολύ ευρία πλειοψηφία και χαίρομαι που μπορούμε να συζητούμε πλέον με το Συμβούλιο, να ευχαριστήσω ήρθαμε παρέοδο όλους τους κοιόδης, και όλη την ομάδα μπορούμε να πάμε απευθείας σε τριμερή διάλογο. Also Προτείνεται λοιπόν να προχωρήσουμε κατευθείαν στον τριμερή διάλογο. Δηλαδή να ξεκινήσουμε αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Μόλις εγκρίναμε την εντολή για αυτό. Η ομάδα διαπραγμάτευση. Ε, θα έχει εμένα πρόεδρα, την κυρία Σαρνέ ε, ω εισηγήτρια και μετά έχουμε του κοιόδους εισηγητέ. Herrn Saradiel, Frau Keller, Herrn Scholz und Herrn Borelli und ein Mitglied von καθώς ε, και ένα μέλος του ΙΕΝΕΦ e εφόσον το επιθυμείτε. Όποιος ε, συμφωνεί παρακαλώ να το δηλώσει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν, αρχή της ψηφοφορίας. Und die Abstimmung ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας. Σχεδόν ομόφωνα. Κάθε επιτυχία στις ε, διαπραγματεύσεις σας εύχομαι, ε, κυρία Ντεσαρνές. Προχωράμε στο σημείο 8 της σημερινής διάταξης. Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών. Έχουμε εδώ καταρχάς την συμβαστική προπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, προφορική τροπολογία του, της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται ηλεκτρονική επαλήθευση Τροπολογία 21, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 5, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αρχή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 29. Λήξη της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και ψηφίζουμε την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Έμα, συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Γνωμοδότηση για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών. στον τομέα της ενέργειας. Ο κύριος Μπένσεν είναι, γνωμοδο... είναι συντάκτης της Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά υπέρ υπέρ. Εγκρίνεται η 41 λοιπόν. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές ε, ας ελέγξουμε 48 αρχή της ψηφοφορίας Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μάλλον ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 65 αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κα... Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε μαζί την 68 μέχρι την 76 68 έως 76. Προτείνεται να ψηφίσουμε μαζί την 68 έως την 76. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Από ό,τι φαίνεται όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί τις τροπολογίες 68 έως και 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική απαλήθευση. 78 αρχή της ψηφοφορίας λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε μαζί τις 9 έως 12. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι. 9 έως 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε την τροπολογία όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά αρχή της ψηφοφορίας ist geschlossen. Λήξη της ψηφοφορίας με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες σήμερα. Όποιος θα ήθελε να εγκαταλείψει την αίθουσα, παρακαλώ ησυχία. Punkt 10 Σημείο 10 παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων μετά την, την προηγούμενη συνεδρίαση. Σας παρακαλώ ησυχία. Είχαμε λοιπόν ε, την ομάδα για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες 1η ε, Σεπτεμβρίου. Δεν ήμουν παρόν, αλλά η Μαρίσα με αντικατέστησε. Μήπως θα μπορούσε να μας μιλήσεις για την ε, ομάδα παρακολούθησης. you like to say something about the... No. Sorry, I was still distracted by everybody <laughs> coming in and out. Ε, συγγνώμη, μου αποσπούσαν την προσοχή όσοι μπαίνουν και βγαίνουν. Ε, θέλετε να μιλήσω για την ομάδα παρακολούθησης. Νομίζω ότι προχωρούν τα πράγματα όπως αναμέναμε και ότι είχαμε επικοδομητικές συζητήσεις ε, με τον κύριο διαπραγματευτή για την TTIP. Ε, δεν έχω να σας πω κάτι ουσιαστικό. Νομίζω ότι η ομάδα παρακολούθησης διευκρινίζει σημαντικά θέματα των Ευρωβουλευτών και νομίζω ότι θα ε, συμβάλλει στην ε, πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί αρχές Οκτωβρίου, νομίζω. Ναι. Τίσα. 7 Σεπτεμβρίου είχαμε συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης ε, με τον κύριο Κίνα, που είναι ο κύριος διαπραγματευτής. Μετά τον 19ο γύρο, όπου προείδρευε η Αυστραλία. Χωρίς πάλι συγκλονιστικά νέα. Αυτές ήταν λοιπόν οι μόνες ομάδες παρακολούθησης που είχαμε. Προχωράμε στο σημείο 11. Έκθεση της κοινή αποστολής ίντα και ανάπτυξης ε, στην διάσκεψη της UNCTAD στο Ναϊρόμπι Δύο θέματα είχαμε εδώ, την συζήτηση για νέα εντολή της UNCTAD που συνδέεται και με το θέμα των μελετών σχετικά με την προβληματική των χρεών και τον πολιτικό ρόλο της UNCTAD, κατά πώς θα πρέπει να ενισχυθεί. Στις διαπραγματεύσεις αυτές συμμετείχαμε εμέσως ε, αφού είχαμε ανταλλαγές απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, υπήρχαν διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις που εξέταζαν διάφορες πτυχές ε, του παγκοσμίου εμπορίου. Ιδιαίτερα ενδιαφερθήκαμε για το Παγκόσμιο Φόρουμ Επενδύσεων Είχα τη δυνατότητα να κάνω μια ομιλία πολύ βασική πάνω στα βασικά θέματα, αλλά επίσης με πολύ ενδιαφέρον ε, παρουσιάσαμε το σύστημα που έχουμε μαζί με τους Καναδούς ε, για το δικαστήριο επενδυτών και λάβαμε πολύ ενδιαφέρουσες αντιδράσεις από τα άλλα κράτη-μέλη. συμφωνήσαμε να συνεχιστεί η συζήτηση. Ιδιαίτερα από τρίτες χώρες τέθηκε το ερώτημα πώς θα διατεθεί το απαραίτητο δυναμικό για την πληρωμή και για την εκπαίδευση, την κατάρτιση των δικαστών. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Παράλληλα είχαμε μια σειρά συνομιλιών και με την Κένια σχετικά με την υπογραφή της ε, εμπορικής ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Και όπως είπαμε στις 20 Σεπτεμβρίου επικύρωσε το Κοινοβούλιο τη συμφωνία αυτή. Κατά τα άλλα έχετε μπροστά σας την έκθεση. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Όχι. Προχωράμε στο σημείο 12. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία. Και δίνω το λόγο κατευθείαν στον εισηγητή Εμμανουέλ Μορέλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη είχαμε εντελεχή συζήτηση τη Ιορδανίας στην προηγούμενη συνεδρία της ΣΥΝΤΑ και ήμασταν ομόφωνοι σχεδόν και για τη διάγνωση και για τις λύσεις προκειμένου να επιληθούν μια σειρά προβλήματα. Ευελιξία των κανόνων προέλευσης ε, και μια ταχεία χρηματοοικονομική στήριξη ε, γενναιόδορη θα έλεγα, εκτός από ταχεία. Ε, μαζί με την Κομισιόν υπήρξε συμφωνία για το μακροοικονομικό στρατηγικό πλαίσιο για τη σχέση με την Ιορδανία οι διαπραγματεύσει ε, για μια τέτοια συμφωνία ε, ε, τίθενται σε στενό ορίζοντα, σε άμεσο ορίζοντα και οι διαπραγματευτές όπως και για την Τινησία λένε ότι θα έχουμε μια ασυμμετρική προσέγγιση και αυτό επιθυμούμε. Για την Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών λοιπόν υπάρχουν κάποιες τεχνικές τροποποιήσεις ε, έναντι μιας κλασικής συμβάσεως που προτείνει η Κομισιόν. Ε, δεν είναι κάτι που θα συγκινούσε τα πλήθη, αλλά εν πάση είναι ε, σημαντικό να φτάσουμε σε μια συμφωνία και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ευέλικτη και ευφυής στην διαπραγματευσή της. Χρειάζεται όμως μια ταχύτατη ενίσχυση, επαναλαμβάνω, και χαίρομαι και η δουλειά της Επιτροπής ΑΦΕΤ επ' αυτού. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα τοποθετηθεί στις επόμενες ημέρες, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μας παρακολουθεί στην πορεία που θα χαράξουμε από κοινού. Θα πρέπει λοιπόν να παράσχουμε μία ενίσχυση για τις χρηματοοικονομικές ε, ε, ανάγκες 16-17 στην Ιορδανία είχα μιλήσει με αρκετούς συναδέλφους ε, και με πιο ειδικού επί των ε, θεμάτων από το ΑΜΑΝ και κάτι που αφορά και στους κοιόδης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιαδήποτε αύξηση θα ήταν προς το συμφέρον των εταίρων ε, από την Ιορδανία και θα πρέπει να έχουμε, εν περιπτώσει, περιθώριο προϋπολογισμού για να μπορούμε να κάνουμε την οποιαδήποτε προσέγγιση. Δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει και στα πλαίσια του, της συνάντησης του Λονδίνου. Επομένως, ε, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω την άποψη των συναδελφών από αυτού, επί του περιθωρίου αυτού. Αλλά εφόσον ήμασταν ομόφωνοι επί της διαγνώσεως, άλλο τόσο ομόφωνοι πρέπει να είμαστε και επί των προτάσεων που σας συστήνω να υιοθετήσουμε. Ευχαριστούμε αγαπητέ Εμμανουέλ. Ε, ο Ντάνιελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Εξ ονόματος του συναδέλφου Τσίκου και του Έλκε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Καλό θα ήταν πράγματι να υποβάλουμε μια ενιαία πρόταση προκειμένου να ενισχυθεί η χώρα αυτή προς την οποία έχουμε σημαντικό ενδιαφέρον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Μορέλ έχει δίκιο επί των πάντων όλων των παρατηρήσεών τους. Υπάρχει το θέμα των προσφύγων, υπάρχει το θέμα του τουρισμού που απουσιάζει δηλαδή πλέον. Έχουμε ένα περιφερειακό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν εξομαλύνεται, ιδιαίτερα αν δούμε τους βομβαρδισμούς αυτή τη στιγμή στο Χαλέπι. Ε, έχουμε επίγουσα ανάγκη ενίσχυσης προς τη χώρα αυτή καλό θα ήταν η Επιτροπή από καιρού καιρών να ε, τηρεί τι δεσμεύσει τη. Ε, είχε πει ότι η Ορδανία δεν θα ήταν, δεν θα υπήρχε εμπόδιο, ε, εν πάση περιπτώσει, προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα επανέρχεται, τέλο πάντων εγώ υποστηρίζω απολύτω τον εισηγητή και τι οποιαδήποτε τροπολογίε υποβάλλει προκειμένου να δοθούν αυτές οι ενισχύσεις ταχεία, ταχαίως θα χρειαστεί κατάλληλη ενίσχυση και μάλιστα ταχύτατα, διότι δεν έχει νόημα αυτή η όλη προσπάθεια. Ο Χέλμον. Ε, και ο κύριος Σόλτς. Πρόεδρε. Από πλευράς του δικού μας σκιώδου συγκητή, ήθελα να πω κάτι που δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα. Όλοι αντιλαμβάνομαι πόσο έχει χτυπηθεί η χώρα από τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας και από το προσφυγικό. Οπωσδήποτε και υπάρχουν ελληνικέ συνέπειε όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και ακριβώς όπως και ο εισηγητής και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ιορδανία. Η βοήθειά μας είναι αναγκαία, άρα χρειάζεται η μαγροοικονομική συνδρομή. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά εν λόγω έργα. Θα πρέπει να ε, γίνει με ρυθμό ανάλογο του επίγοντος της καταστάσεως. Έχουμε άλλωστε το άρθρο 3 παράγραφος 2. Και άρα θα πρέπει η μακροοικονομική συνδρομή έτσι να χορηγηθεί στην Ιορδανία σε σχέση και με τα ανθρώπινα δικαιώματα μια που δεν υπάρχει ελευθερία τύπου δεν υπάρχει κανένας είδους ουσιαστική αντιπολίτευση Ακούσαμε πρόσφατα βέβαια την πολύ καλή ομιλία του, στο, του Βασιλέα στο Στρασβούργο σχετικά με τους πρόσφυγες, αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε τα άλλα θέματα. Αυτές λοιπόν ε, είναι οι σκέψεις μας, τις οποίες θέλουμε να υποβάλουμε και στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας μιλώ για του συναδέλφου Λούνας, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί. Θα ήθελα όμως να αναφέρει ότι η πολιτική μας ομάδα να γνωρίζει όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η, η Ορδανία όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων από τη Συρία. Και αναγνωρίζουμε επίση όλα τα προβλήματα που προκύπτουν αυτές τις προσπάθειες, οπότε και εμείς συμφωνούμε με τη χορήγηση της ε, οικονομικής ενίσχυσης και θεωρούμε ότι βέβαια θα πρέπει η προϋπόθεση να είναι η ορθή αξιοποίηση των πόρων που θα λάβει η χώρα. Ο κ. Λούνες επίσης μου ανέφερε το εξή. Ο εισηγητής του είπε κατά πόσον ε, θέλει να προσυπογράψει μια τροπολογία γιατί έχουμε αυτά τα 200 έως 350 εκατομμύρια ευρώ αλλά προ το παρόν είπαμε ότι επιφυλασσόμαστε και δεν θα προσυγουράσουμε αυτή την τροπολογία. Αλλά θα το σκεφτούμε. Επίσης, όσον αφορά την τροπολογία, περιμένουμε να μας ενημερώσει για το τι γίνεται ε, η Επιτροπή για τις ανάγκες τη χρηματοδότηση. Οπότε όταν ενημερωθούμε θα λάβουμε και την τελική μας απόφαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ιορδανία, γιατί κάτι. Αγαπητέ Πρόεδρε, προχωρήσατε τόσο γρήγορα την με στι διάταξη που οι συνάδελφοι για τα χρηματοοικονομικά δεν ήρθαν ακόμα αλλά όλα σου άκουσα θα τα σημειώσω και θα τους τα διαβιβάσω. Um... Όπως πάντα, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Εμμανουέλ. Δεν κατάλαβα καλά, τέλο πάντων θα πούμε άλλη ώρα με την Ευρωπαϊκή Οτροπία. Ευχαριστώ για όλα αυτά που ρώτησαν οι συνάδελφοι, οι θεμητέ ερωτήσει και ο κύριο Σόλτ σωστά τα λέω και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Επίση, ευχαριστώ του περισσότερου αδέλφου οι οποίοι είπαν ότι συμφωνούν με την πρότασή μου να αυξήσουμε το σχετικό ποσό. Δεν είναι θέμα μαξιμαλισμού. Είναι το ότι τόσα χρειάζονται. Το είπε και η κυρία Ντεσσαρνέ, αλλά το είπαν και άλλοι. Πρόκειται μια χώρα που έχει πάρα πολλέ δυσκολίε. Οπότε θεωρώ ότι η Ένωση που θέλει να βοηθήσει τις χώρες της περιοχής αυτής θα πρέπει τα λόγια να τα κάνει έργα. Ε, γι' αυτό και κατέβασα τη σχετική τροπολογία. Ε, ευχαριστώ για την ποιότητα της συζήτηση και θα τα πούμε την Κομισιόν. Ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε. das soll auch so sein. Ähm, ja, grundsätzlich ist Γενικά, θα πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτήν την πρόταση. Διότι η Ιορδανία φέρει σημαντικό βάρος και θέλουμε στον, ε, να, να τη στηρίξουμε σε θέματα που επηρεάζουν τον ε, τουρισμό και άλλες πηχές. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να βλέπουμε και την, ε, τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Βλέπουμε προσέλευση πολλών Σουνιτών που μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση. Θα πρότεινα λοιπόν μαζί με την υποστήριξη να έχουμε και παρακολούθηση της πολιτικής κατάστασης ώστε να μην μας ξεφύγει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής τα κατέγραψε όλα. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Σεπτεμβρίου. 7 η ώρα το βράδυ. Και η ψηφοφορία στην Ίντα θα πραγματοποιηθεί 12-13 Οκτωβρίου στην επόμενη συνεδρίαση δηλαδή της Ίντα. Και περνάμε στο σημείο 13. Προσχώρηση στη Συμφωνία Εμπορίου της Κολομβίας και του Περού ε, από τον Ισημερινό. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 17 Ιουλίου. 2014. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα το θέμα αυτό. Στείλαμε τον Μάρτιο του 2016 μία αποστολή ad hoc στον Ισημερινό και ακολούθησε ψήφισμα. Και προσπαθήσαμε να ασκήσουμε πίεση για ε, σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε ο Ισημερινός να μην έχει πρόβλημα ε, στο κενό ανάμεσα στην συμφωνία και τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πολλές συζητήσεις. και με το Συμβούλιο και την Κομισιόν και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χέλμουτ Σόλς. Ο οποίος θα μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήδη αναφέρατε τα πιο σημαντικά θέματα εδώ. Σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία αυτή, δηλαδή θα πρέπει να βρούμε την μία λύση εντός του ετούς, εντός του 16. Διότι από του χρόνου ο Ισημερινός θα χάσει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα για τη χώρα αυτή και για όλους εκείνους που εργάζονται στους διαφορετικούς οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε δηλαδή την συνεχιζόμενη πρόοδο για τα δημοκρατικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα και για να είμαστε σαφείς τους τελευταίους μήνες για να μην πω χρόνια ήμασταν σε επαφή με την Επιτροπή και τις προεδρίες σχετικά με την ολοκλήρωση αυτού του πρωτοκόλλου προσχώρησης και σύμφωνα και με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου όπου είχαμε ήδη σηματοδοτήσει ποιες θα, πρέπει, ποιες θα έπρεπε να είναι κατευθυντήριες γραμμές για την προσχώρηση. Έχουμε υπογραμμίσει λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες τυχές και δυσκολίες και πέραν αυτών έχουμε προσθέσει και το θέμα των επιπτώσεων του σεισμού την Άνοιξη φέτος που έπληξε τον Ισημερινό και που δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες παρά πέραν μάλλον των ήδη υφισταμένων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Θα πρότεινα λοιπόν μια θετική στάση του Κοινοβουλίου προς την επικύρωση της συμφωνίας αλλά βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε την επίσημη διαδικασία μετά την υιοθέτηση του Συμβουλίου. Και βεβαίω πάντα πρέπει να εμένουμε στις δημοκρατικές επιταγές του Κοινοβουλίου να ελέγχουμε συνεχώς ποιο είναι το πλαίσιο της συμφωνίας, τι επιπτώσεις θα έχει επί των πολιτών και των 28 κρατών μελών. Όπως και επί των επιχειρήσεων, όπως και επί των κοινωνικών εταίρων στην άλλη χώρα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε στα πλαίσια κάθε συμφωνίας με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη θέση μας αυτή τη στιγμή. Και ξέρουμε ότι έχουμε πρόσθετες προκλήσεις. Είχαμε και την πληροφορία για τις ε, ρήτρες διασφάλισης που είναι ένα αντίστοιχο Παράδειγμα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη γεωργία, για άλλους οικονομικούς ε, τομείς και της χώρας της ενδιαφερόμενης ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, συνάδελφοι, θα ζητούσα όταν υποβάλλω το σχέδιο έκθεσης να μπορέσουμε στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα να τη συζητήσουμε και να την ψηφίσουμε ώστε να έχουμε ολοκληρώσει την όλη διαδικασία της επικύρωσης μέχρι το Δεκέμβριο με τις Ολομέλειες. Δηλαδή πριν από την ε, συνάντηση στις 29 Νοεμβρίου θα πρέπει να ελέγξουμε την έκθεση. Είναι σύντομη η προθεσμία ενόψης της ολομέλειας του Δεκεμβρίου, αλλά ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου ότι εδώ θα πρέπει να εξεύρουμε μια ισορροπία και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για εκείνους τη σημερινή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχουν οι σκιώδεις. Συνάδελφοι, ο Σφίσα σκιώδη ε, δεν μπορεί να είναι παρόν σήμερα, γι' αυτό θα ήθελα να διαβάσω τις παρατηρήσεις του. Όσον αφορά τη διαδικασία, το ΕΛΚ ε, διατηρεί τη δέσμευσή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προσχώρηση του Ισημερινού μέχρι το τέλος της χρονιάς ε, και με την ε, διότι το 2014 εκπνέει το σύστημα GSP Plus και θα πρέπει να στηρίξουμε την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νότια Αμερική. Ε, κάτι, για το οποίο αποτελεί, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητο ε, η προσχώρηση του η σημερινού. Και επίσης θα θέλαμε να υπάρχει συνένεση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά το σχέδιο δράσης, ε, έχουμε διαβάσει το σχέδιο δράσης για τον Ισημερινό ε, σχετικά με ε, ισχύοντα και μελλοντικά νομοθετικά μέτρα και υπάρχει ψήφισμα του 2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την διαδικασία ε, και μετά την θέση σε ισχύ της συμφωνίας στο πνεύμα ε, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης όπως κάνουμε και με τους άλλους εταίρους, ε, την Κολομβία και το Περού. Επίσης όσον αφορά το TBT και το SPS σημειώνουμε τις καλές εξελίξεις αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζεται άμεση δράση από πλευρά του Ισημερινού για την άρση των ποσοστώσεων για τις εισαγωγές αυτοκινήτων που αντίκυνται στις υποχρεώσεις ε, του Ισημερινού στο πλαίσιο του ΠΟΕ και περιμένουμε σημαντικά βήματα σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών μπορώ να πω ότι και εμείς ενδιαφερόμαστε για ολοκλήρωση της προσχώρησης για να μην υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τον Ισημερινό. Και θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τον διάλογο με τον Ισημερινό. Χρειάζονται λοιπόν ακόμα κάποια πράγματα. Και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. και όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της βιωσιμότητας. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα αποφασίσει το Συμβούλιο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο να ολοκληρώσουμε την προσχώρηση. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα στηρίζαμε το θέμα αυτό και ακόμα περισσότερο στηρίζουμε το θέμα αυτό τώρα που βλέπουμε ότι το γενικό κλίμα για το ελεύθερο εμπόριο και τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου επιδεινώνεται παγκοσμίω. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσει η προσχώρηση του Εκβαδόρ σε αυτήν την εμπορική συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Πιστεύουμε ότι θα ωφελήσει την Ευρώπη, τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, διότι ανοίγουν νέες αγορές για σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία ή τα αλκοολούχα ποτά. Πιστεύουμε επίσης ότι η συμφωνία αυτή θα ωφελήσει και το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό, διότι θα αποτελέσει κινητήρια για την οικονομική ανάπτυξη και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, ιδιαίτερα της ακραίας φτώχειας σε υπαίθριες περιοχές. Να τονίσω επίσης ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει σημαντική αναπτυξιακή πτυχή στην προσχώρηση του Ισημερινού, καθότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σημαντικότερη αγορά για τις μη πετρελαϊκές εξαγωγές ε, ε, ε, του Ισημερινού, καθώς και η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ισημερινού. Χαιρόμαστε που έχει επιταχυνθεί η διαδικασία και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να επικυρωθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς κάτι που θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε το κενό καθώς και τη ε, ε, διατάραξη των εμπορικών ροών. Μία τελευταία παρατήρηση και μία ερώτηση προς τον εισηγητή ή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την Κολομβία και το Περού. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δυσκολίες από την πλευρά τους. Ε, θα ήταν χρήσιμο να το γνωρίζουμε. Όπως και να έχει, προσλέπω στην καλή συνεργασία με τον εισηγητή. Και τον στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Να δώσω το λόγο τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Γιώργενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα με κατηγορήσουμε και εμείς. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό του να προσχωρήσει ταχύω ο σημερινό στην εμπορική συμφωνία ΕΕ γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό ότι εδώ πέρα υπάρχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή σα προ τούτο. Ε, Επίση, να σα αναφέρουμε ότι θέλουμε να συγχαρούμε τη χώρα για τι ε, προσπάθειε που έχει καταβάλει, για το έργο που έχει επιτελέσει τώρα τελευταίο, τόσο ώστε να επιληθούν τα προβλήματα τα σχετικά με το εμπόριο. Προετοιμάζονται για την προσχώρηση. Είναι αξιόλογες οι προσπάθειες. Πρέπει να συνεργαστούμε. Πάντως, ακόμα χρειάζεται δουλειά σε διάφορα μέτωπα. Ιδίως όσον αφορά τις για τα αυτοκίνητα. Μας προβληματίζει το θέμα και έχουμε πιέσει το σημερινό να μας ε, ε, βεβαιώσει ότι θα καταργηθούν αυτές οι ποσοστώσεις. Να το τονίσουμε αυτό. Τέλος. Όσον αφορά το πώς έχουν τα πράγματα με Κολομβία και Περού, είναι οικοδομητικές οι σχέσεις μας, συνεργαζόμαστε για τα τεχνικά θέματα και οι ενδείξεις είναι ότι και η Κολομβία θα βελτιώσει τις επιδόσεις της και θα είναι έτοιμη για προσχώρηση όσον αφορά το πρωτόκολλο όποτε ορίσει και αποφασίσει το Συμβούλιο. Βέβαια, θα δούμε τελικά τι θα πει, πούν και οι σε αυτές τις χώρες Κολομβία και πέρα πρόεδρος. Έχουμε τίποτε νέα από πλευρά Συμβουλίου πώς ε, προχωρούν τα θέματα με την προθεσμία της 11ης 11ου. Το Συμβούλιο. Ή μάλλον η Επιτροπή. Από ό,τι γνωρίζουμε ε, ισχύει ακόμη. Σου έχουμε πει να επιταχύνουν τους ρυθμούς να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την απόφαση της υπογραφής της συμφωνίας. Του λέμε για Οκτώβριο, αυτή οπότε μαζί όμω δεν έχει αλλάξει η προθεσμία της 11 η Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος, πολύ καλά. Ε. Και δίνει το λόγο στον κύριο Σόλτσο. Ελπίζω ότι αυτά που είπε στο τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιηθούν. Θα πραγματοποιηθούν δηλαδή και δεν θα φρενάρει άλλο τη διαδικασία και τις εξελίξεις του Συμβουλίου. Και είναι και ο ίδιος ο πρόεδρος Προσπαθούμε σε στενή συνεργασία με την Προεδρία να επηρεάσουμε τις ε, διαδικασίες για να υπογραφεί το πρωτόκολλο. Και βέβαια η χώρα, ο έχει παρουσιάσει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα που απηχεί τις προσπαθίες τους. Άρα είναι θέμα ανάπτυξη της χώρας. Και πρέπει να δούμε πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα που ανέφεραν σήμερα διάφοροι συνάδελφοι. Και πρέπει επίσης να ξεβρεθούν λύσεις και για άλλα οικονομικά προβλήματα που αφορούν το Εκουαδόρ και την οικονομία του. Ας πούμε το σωσίγιο πληρωμών, τις σχετικές ε, ρήτρες θα πρέπει να, να καταστεί βέβαια ότι όλα θα γίνουν όπως προβλέπονται στα πλαίσια όσων προβλέπει ο ΠΟΕ ε, που θα πρέπει βέβαια να τηρήσει τα υπεσχημένα και η διεθνή κοινότητα αντιστοίχως και να βρεθούν οι απαντήσεις για τα προβλήματα που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίω και εγώ θεωρώ ότι θα τηρήσετε επισχυμένα το Συμβούλιο και θα τηρηθεί αυτή η προθεσμία της 11ης Νοεμβρίου για το πρωτόκολλο. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο βέβαια και θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, τότε όλοι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι υπόλοιπες χώρες, ιδίως το Εκουαδόρ. Άρα θα πρέπει να εφαρμοστεί ότι προβλέπει για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και οπότε και εμείς από πλευρά Συνοτικής Αριστεράς θεωρούμε ότι πάνε τα πράγματα καλά. Αν όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αν δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία έχουν συζητήσει τόσα, τόσους μήνες, τόσα χρόνια, ε, τότε είναι θέμα απώλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέμα ε, απουσίας δικής μεταχείρισης των χρόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ας προσεγγίσουμε σωστά το θέμα όλες οι πολιτικές ομάδες. Και ας ελπίσουμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και πλευρά των 28 κρατών μελών. Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από πλευρά Συμβουλίου. Και εμείς θα συνεργήσουμε όσο γίνεται γρήγορότερα. Θέλουμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητούν αυτά στην επόμενη συνδέσή μας ως έκθεση και ελπίζουμε ότι θα έχει αποφασίσει το Συμβούλιο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου και εμείς θα εγκρίνουμε την έκθεση στη συνεδρίαση του 29 Νοεμβρίου και το κείμενο θα κατέβει στην ε, Ολομέλεια του Δεκεμβρίου το τελευταίο. Είναι η συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία. Άρα, θα καλούσα εκτός το Προεδρείο της Επιτροπής για τη σχέση με την Τουρκία, τα μέλη, τους βοηθούς που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Όλους τους υπολείπους δηλαδή να αποχωρήσουν παρακαλώ. κανείς